Herr Präsident! Guten Tag. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ich erkläre die am 27. November Κηρύττω την ε, επανάληψη της Συνόδου Ολομέλειας που διακόπησε στις 27 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι μια βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ναι. Τουρκία είναι μια χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση